Dear colleagues, good morning. Καλημέρα σε αγαπητοί συνάδελφοι. Παρόλο που δεν είναι κατάμεστη αίθουσα ακόμη, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να προτανθώ πρώτα στα μέλη τη ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Καταρχήν, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει, μήπω. Όχι, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η αυριανή συνεδρίαση των συντονιστών θα αρχίσει αύριο στι 10 παρατέταρτο και όχι στι 9.30 όπω αρχικά είχαμε προγραμματίσει. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις του Προέδρου, το σημείο 2 δηλαδή. Και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 3. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ το συμπρόεδρο για το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, τον κύριο Κλοντ Μωράες, που όπως γνωρίζετε είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Γιατί το σημείο 3 προβλέπει συζήτηση σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Λίμπε και Γιούρη. Θα ακούσουμε λοιπόν από κοινού την παρουσίαση της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση των Δικαστών για το 2015. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Κλοντ Μωράς. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συμπρόεδρε Πάβελ και αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έχω την ευκαιρία να συμπροεδρεύσω στη συνεδρία σε αυτή με τον Παύλ Σφόμποντα και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων για την κατάρτιση των δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και για την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, τη ΛΥΜΠΕ. Και ακριβώς πριν την έναρξη της συνεδρίασης ε, συζητούσαμε πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε με την Επιτροπή Γιούρι το θέμα αυτό. Και εγώ και ο προκατοχός μου, ο κύριος Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ, φροντίσαμε να θέσουμε αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα της συνεργασίας των δύο επιτροπών. Οπότε μετά το, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1999 αναγάγαμε την κατάρτιση των δικαστών σε βασικό ζήτημα της συνεργασίας στα θέματα ποινικού δικαίου. Και οι δύο επιτροπές, Γιούρι και Λίμπε, ασχολούνται με θέματα ε, ποινικού δικαίου και η συνεργασία μας ήταν ανέκαθεν πολύ σημαντική. Και μάλιστα και η κυρία Κοντρίσκα και η κυρία Τσενίτση, αντιπρόεδροι, πρόσφατα ολοκλήρωσαν μια σχετική έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ε, για τη αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα. Η αμοιβαία αναγνώριση, μάλιστα, στο θέμα αυτό προποθέτει εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, Ευρωπαίων δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων. Κάτι που προποθέτει εξοικείωση με τα άλλα νομικά συστήματα και την δημιουργία μιας ε, ευρωπαϊκής ε, νομικής κουλτούρας. Θέλει χρόνο αυτό. Για να δημιουργηθεί μια τέτοια κουλτούρα είχαμε και σχετικό ψήφισμα τον Ιούνιο του 2010 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρμοδιότητα για την ε, πρόθεση της κατάρτισης ε, των δικαστών και ε, υπάλληλων των δικαστηρίων σε τέτοια θέματα δικαστική συνδρομή. και είναι απαραίτητο στοιχείο για να υλοποιηθούν και τα οι προτεραιότητες και οι στόχοι του ψηφίσματός μας. Ε, και μάλιστα έχουμε στα θέματα της ε, Ευρωπαϊκής της αστυνομικής συνεργασίας και της ε, δικαστικής συνδρομής σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης αρμοδιότητα κοινοτική. Αυτά είναι τα προκαταρκτικά μου σχόλια και μετά από αυτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο τον κύριο Σφόποντα. Με κάθε σεβασμό και προς εσένα θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε εμείς εδώ οι δύο οι πρωταγωνιστές αυτής της συνεδρίας, αλλά κυρία Άστολα που έχει αναλάβει πρόσφατα Γενική Διευθύντρια για θέματα δικαιοσύνης και δικαιωμάτων των καταναλωτών στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχαρητήρια κυρία μου για το διορισμό σας και να σας δώσω το λόγο για την ενημέρωση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους Πρόεδρους ε, της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων, τον κύριο Σπόμποντα και των Πολιτικών Ελευθεριών, τον κύριο Κλοντ Μωράες, για την ευκαιρία που μου δίνουν σήμερα να σας ε, παρουσιάσω τα τελευταία απορίσματα και τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση Δικαστών. Αυτή μάλιστα είναι η παρθενική μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και Προστασία των Καταναλωτών, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χαίρομαι γιατί θα συζητήσουμε ένα θεμελιώδη ζήτημα που αφορά όλους μας. Πώς θα εξασφαλίσουμε οι επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης ε, να γνωρίζουν πώς θα εφαρμόσουν σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, το Ενωσιακό Δίκαιο. Κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο. Χρήζει συνεχούς προσπάθειας. Και μάλιστα η νομοθεσία μας εφαρμόζεται εμπράκτως μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά. Η κατάρτιση λοιπόν των δικαστών είναι θεμελιώδους σημασία για την ε, ε, εύρυθμη συνεργασία σε συνοριακά θέματα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνη. Η κατάρτιση μάλιστα αυτή δίνει ζωή και ουσία και περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη. εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίε στον τομέα της δικαιοσύνη ε, που συμμετέχουν στις διάφορες ε, δίκε ε, ή στην εκτέλεσή του, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη ενημέρωση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για το ενωσιακό δίκαιο και μάλιστα επικαιροποιημένη συμφωνούμε και στηρίζουμε αυτή την κατάρτιση των δικαστών και των υπαλλήλων του δικαστικού συστήματος. Και μάλιστα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012 εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013 και 2014 και το σχετικό πρόγραμμα συνέβαλε στην ποιοτική βελτίωση της κατάρτισης ε, των δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων. Και μάλιστα τα δικά σας ψηφίσματα για την κατάρτιση αυτή άλλαξε το τοπίο της ε, κατάρτισης των ε, δικαστών, δικηγόρων και ε, εισαγγελέων. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψε. Μάλιστα θα σας παρουσιάσω σήμερα τις πρόσφατες εξελίξεις ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Δικαστική Κατάρτιση, ιδιαίτερα στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Επίσης θα σας ενημερώσω για την κατάσταση του επιμέρους κρατημέλη πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ε, ε, του φιλόδοξου στόχου της ε, κατάρτισης 700.000 ε, υπαλλήλων στον τομέα της δικαιοσύνης. Έχουμε ένα μηχανισμό μάλιστα υποβολής εκθέσεων από αρμοδίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι βελτιώνουμε και επικαιροποιούμε τα στοιχεία με βάση τις εμπειρίες που συγκεντρώνουμε. Στόχος μας είναι ένας μηχανισμός που θα μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε που συντελείται πρόοδος και που υπάρχουν αδυναμίες, χωρίς όμως να πολλαπλασιάζουμε το διοικητικό φόρτο. Σε ό,τι αφορά τις τάσεις και που βρισκόμαστε σήμερα. Τα χαρμόσυνα μαντάτα είναι ότι οι καλές τάσεις του παρελθόντος για την Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση διατηρούνται. Το 2014 είχαμε πάνω από 132.000 απασχολούμενους στο δικαστικό που ε, παρακολούθησαν μια κατάρτιση, δηλαδή 13.000 ε, επιπλέον σε σχέση με το 2013. Και μάλιστα από το 2011, την τετραετία που ακολούθησε, σχεδόν υλοποιήσαμε το μισό μας στόχο ε, από το ορόσημο που έχουμε δώσει θέση για το 2020. Και αν διατηρηθεί το παρόν επίπεδο συμμετοχής και στο μέλλον μέχρι το 2020 όχι μόνο θα υλοποιήσουμε αλλά και θα υπερβούμε το στόχο μας για την κατάρτιση των δικαστών και των υπαλλήλων στο τομέα της δικαιοσύνης. Τώρα, κάποιες καινοτομίες. Το 2014 το επίπεδο συμμετοχής έχει αυξηθεί για όλα τα επαγγέλματα. Δικαστές και εισαγγελείς φυσικά είναι στην πρώτη γραμμή, φυσικά εν μέρει χάρη στην την υποστήριξη του δικτύου δικαστικής κατάρτισης που ε, χρηματοδοτείται από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τους συμβολογράφους είχαμε μεγάλη, συμμετοχή της, ε, μεγάλη αύξηση συμμετοχής από 21% στο 31% ε, επαγγελματιών που καταρτίστηκαν στο ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με το 2013. Και μάλιστα εποφελούνται από σημαντικέ κοινοτικέ ε, επιδοτήσει για κατάρτιση ό,τι αφορά θέματα κληρονομικής διαδοχής, η αναγνώριση και εφαρμογή των αποφάσεων σε εμπορικά και ζητήματα του αστικού δικαίου. Φυσικά, η χρηματική υποστήριξη που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την, την ε, αφύπνιση των δικαστών για το πόσο σημαντική είναι η ε, ανάγκη αυτή της κατάρτιση. Επίσης, σε ό,τι αφορά του δικηγόρου έγινε μια κατανομή που δίνει μια πολύ μερική εικόνα, γιατί ακόμη μας λείπουν στοιχεία, κυρίως ε, από τους ε, ε, ιδιωτικού παρόχους κατάρτιση. Βέβαια, είναι δύσκολο και για τους δικηγορικούς συλλόγους να εντοπίσουν αυτούς τους παρόχους για να αποκομίσουν στοιχεία για το επίπεδο κατάρτισης. Σημαντικό εργαλείο για την ε, πρόθεση της προόδου στη συμμετοχή των δικηγόρων είναι να παράσχουμε ε, προσιτές πληροφορίες ότι αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης και θέλουμε να συμπεριλάβουμε και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατάρτισης, ένα ε, επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προϊόν που συμβάλλει ε, μέσω της ε, σχετικής πύλης για την, Ευρωπαϊκή, για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη να βοηθήσει τους επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης ε, να παρακολουθήσουν κατάρτιση μάλιστα σε γλώσσα της επιλογής τους και οπουδήποτε στην Ευρώπη. Βέβαια, λίγη κατάρτιση έχουμε στα θέματα νοσιακού δικαίου για τους δικαστικούς κλητήρες και τους υπαλλήλους των δικαστηρίων. Βέβαια, οι δικαστικοί κλητήρε εφαρμόζουν αυτέ τι ξένες αποφάσεις, τις ε, αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουν την, ε, το ενωσιακό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για την εφαρμογή διασυνοριακά ε, διαθήκων. Γι' αυτό και τον περασμένο Οκτώβριο επικεντρωθήκαμε στην νομική κατάρτιση αυτών ακριβώς των επαγγελματιών της δικαιοσύνης. Είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την σημασία που έχει η ανταλλαγή πρακτικών, των πρακτικών και εμπειριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι επαγγελματίε ζητούν να συνεχιστεί αυτή η κοινοτική υποστήριξη και σε μεγάλο βαθμό θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση των επαρχόντων μαθημάτων ε, κατάρτισης και των, ε, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαστών και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ε, Δημόσιας Διοίκησης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτές οι δομές. Βέβαια με την διάλεξη αυτή αυξήθηκε η εφύπνιση και η ανάγκη συνεργασίας για να προωθηθεί η κατάρτιση και των δικαστικών κλητήρων και των υπαλλήλων των δικαστηρίων. Βέβαια, υπάρχουν διαφορέ ό,τι αφορά το επίπεδο συμμετοχή της κατάρτιση αυτή μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό πάντω οι αρμόδιε αρχέ όχι μόνο να ε, έχουν επίγνωση των αναγκών κατάρτισης, αλλά να προσφέρουν ε, και να παράσχουν και τα κατάλληλα μέσα για την κατάρτιση αυτή. Τώρα, λίγα λόγια για την κοινοτική συνδρομή. Η δικαστική κατάρτιση είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των κρατών μελών, αλλά τα, και της χωρών δικαστών και των ε, πανεπιστημίων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει τη δικαστική κατάρτιση, με βάση δράσεις που στηρίζονται σε τρεις άξονες. Για παράδειγμα, ε, παρέχει οικονομική χρηματοδότηση αυτών των καταρτήσεων, βελτιώνει την ποιότητά τους και εξασφαλίζει ταχύ αντίδραση στις νέες ανάγκες της δικαστικής κατάρτισης. Και να σας πω λίγα λόγια για τις νέες αυτές τάσεις και τους τρεις αυτούς άξονες. Σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη δικαστική κατάρτιση στο μέλλον. Και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της δικαιοσύνης θα δαπανίσει πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επτέτη χρηματοδοτική περίοδο για την δικαστική κατάρτιση. Και ήδη έχει ξεκινήσει η εκταμείευση αυτή. Έχουμε τήσια κονδύλια για το EJTN και θα έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα ειδικά για την ε, δικαστική κατάρτιση. Αρχικά προτάθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2014. Και μάλιστα είδαμε το ζωηρό ενδιαφέρον των επαγγελματιών, γιατί πολλές αιτήσεις κατατέθηκαν και μάλιστα ο προϋπολογισμός αυτός ε, θα δαπανηθεί σε 22 διαφορετικά δικαστικά συστήματα κατάρτισης υψηλή ποιότητας. Επίσης υπάρχουν σχέδια για το αστικό δίκαιο με επίκεντρο την νέα νομοθεσία όπως ε, ο κανονισμός για τις κληρονομικές διαδοχές και την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο και τις προτεραιότητες αυτές, το θέμα των δικονομικών δικαιωμάτων, των ε, θυμάτων ε, των εγκλημάτων ή εναλλακτικέ λύσεις για την, για την κράτηση. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει διαγωνισμό για ένα πρόγραμμα κατάρτισης των υπαλλήλων του δικαστηρίου. Γιατί, επαναλαμβάνω, χρειάζεται αύξηση της κατάρτισης και αυτού και αυτών των επαγγελματιών. Επίσης, ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση για το διαγωνισμό του 2015 για την δικαστική κατάρτιση και επαναλαμβάνω θα δαπανίσουμε τον προπολογισμό μα σε εξαιρετική ποιότητα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, η ποιότητα είναι ακόμη πιο σημαντική από την ποσότητα. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και Δικαιωμάτων των Καταναλωτών φροντίζει να βελτιώνει συνεχώ την, την ποιότητα της κατάρτιση. Πέρυσι είχαμε στενή συνεργασία με ευρύ δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα δικαστική κατάρτιση με αποτέλεσμα να συντάξουμε έναν περιεκτικό οδηγό για τους παρόχους της κατάρτισης, για την καλύτερη προετοιμασία και παρακολούθηση τέτοιων μαθημάτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης. Και καλύπτει όλες τις, όλα τα προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης. Μάλιστα αυτός ο οδηγός θα μεταφραστεί σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες και θα μοιραστεί τα ενδιαφερόμενα επαγγέλματα. Και μάλιστα θα βρείτε τα σχετικά στη δικτυακή πύλη ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Και λίγα λόγια για την άμεση αντίδραση στι αναφιόμενες ανάγκε. Οι ανάγκε τη κατάρτιση δεν είναι σταθερέ. υπάρχουν πάντα καινούργιε ανάγκε που προκύπτουν και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι να τι προλαμβάνουμε και να τι αντιμετωπίζουμε. Και εδώ έρχομαι στι νέε εξελίξει. Το 2015 μετά τι ε, τραγικέ τρομοκρατικέ επιθέσει, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέλαβε δράσει έτσι ώστε οι επαγγελματίε του χώρου τη δικαιοσύνη να μπορούν καλύτερα να αντιμετωπίσουν ε, την ε, τρομοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση μέσω στοχευμένη κατάρτιση. Το δίκτυο κατάρτιση δικαστών ξεκίνησε κάποιε δραστηριότητε για δικαστικού και εισαγγελεί, επικεντρωμένο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία και την πρόληψη και της, ε, την πρόληψη της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Μεταξύ του 2015 και του θα υπάρξουν τέσσερα σεμινάρια για το υπάρχον νομικό πλαίσιο, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Αλλά θα υπάρξει και μια σειρά ανταλλαγών, πρακτικών και εμπειριών με τους επαγγελματίε του κλάδου, έτσι ώστε να μάθει ο ένας από τον άλλον. Αυτά τα είδη κατάρτισης εξακολουθούν να συνεχίζονται. Κάποια πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ πολλά υπασχόμενα και δείχνουν ότι οι επαγγελματίε του κλάδου μπορούν να έχουν μεγάλο ρόλο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Το 2015 το, η δικαστική κατάρτιση ζήτησε, ε, έγιναν προτάσεις ε, για ε, υποβολή θεμάτων αποδόθηκαν αρκετά κονδύλια για την αντιμετώπιση ακριβώ τη τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Η Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνη θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά στι 20 Μαΐου σε μια διάσκεψη μαζί με το Δίκτυο Δικαστική Κατάρτιση. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φυσικά θα προσκληθούν να είναι παρόντε. Ελπίζω να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα για τα μελλοντικά βήματα για την δικαστική κατάρτιση ώστε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και την ριζοσπαστικοποίηση. Κλείνοντα να πω το εξή ε, γιατί είναι κάτι που με ανησυχεί. Η αρχική κατάρτιση για την, ε, νομική, για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους ε, νέους επαγγελματίες. Είδαμε ότι η αρχική κατάρτιση που αποδίδεται για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, είναι, ε, δεν είναι επαρκή για του νέου επαγγελματίε των νομικών επαγγελμάτων. Η εθνική νομοθεσία εμπνέεται προφανώ από την ευρωπαϊκή και είναι σημαντικό να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νομική κουλτούρα ευρωπαϊκή από την αρχή της, από την έναρξη της άσκησης του επαγγέλματο ενός νομικού. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδυαστούν οι προσπάθειες και οι πρακτικές των επαγγελματιών από διάφορες χώρες υπάρχει και το πρόγραμμα IACOS, το οποίο έχει, δημιουργηθεί από το δικαστικό δίκτυο κατάρτιση, που είναι πολύ καλό παράδειγμα για τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών και εισαγγελέων. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές προσπάθειες ε, και από το ε, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης. Το πρόγραμμα όμω το συγκεκριμένο θα χρειαστεί περισσότερη ενίσχυση για να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του, ότι δηλαδή το 2020 όλοι οι νέοι εισαγγελεί και οι δικαστικοί θα έχουν ε, συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγή δύο εβδομάδων. Ακόμη η απορρόφηση του προγράμματος αυτού ε, δεν είναι επαρκής, έχει φτάσει μόλις το, κάτω από το 50% των δικαστικών και εισαγγελέων η ε, συνεργασία λοιπόν με το δικαστικό δίκτυο ε, κατάρτισης είναι, καλό να ενισχυθεί έτσι ώστε να δούμε γιατί το πρόγραμμα IACOS χρησιμοποιείται επαρκώς. Πρέπει επίσης να δούμε πόσο, σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η αρχική κατάρτιση των επαγγελματιών και των νέων ε, δικηγόρων, συμβολιογράφων, δικαστικών υπαλλήλων ε, πρέπει όλοι να γνωρίζουν την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσο πιο νωρί την γνωρίσουν, τόσο πιο καλά θα μπορέσουν να την ενσωματώσουν στην ε, εθνική του νομοθεσία και θα οδηγήσουν σε καλύτερη ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, θα ήθελα να ζητήσω την στήριξή σα για να υποστηρίξετε και εσείς στις δικές σας χώρες και εκλογικές περιφέρειες την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει καλή κατανόηση του ευρωπαϊκού του ευρωπαϊκού δικαίου από την αρχή της έναρξης του επαγγέλματο ε, των ε, νομικών. Αυτό χρειάζεται για να είναι ε, απολύτω αποτελεσματική και απολύτως εφαρμόσιμη η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε η δικαστική κατάρτιση να μείνει ψηλά στην ατζέντα μας. Προσβλέπω φυσικά στην ε, συνέχεια της εργασίας μας έτσι ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα εφαρμόζεται από καλώς κατευθυσμένους ε, νομικούς επαγγελματίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα επιτύχουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την σωστή ολοκλήρωση της του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Thank you very much, madam. Εγώ ευχαριστώ. Πολύτιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις και για απαντήσεις, ελπίζω. Η κυρία Ρέγνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Το παρακολουθούμε το θέμα αυτό εμείς εδώ και καιρό στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ακριβώς αυτοί που θα εφαρμόσουν και θα χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις ε, διατάξεις να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά και έχω κάποια ερωτήματα. Αν δούμε τους πίνακες, υπάρχουν ε, μεγάλες εθνικές διαφορές σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα και την εφαρμογή στην πράξη της, ε, και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης. Ποιες αιτίε υπάρχουν, θα μπορούσατε να μας πείτε εσείς κάτι περισσότερο γι' αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω έχει να κάνει με την διεξαγωγή όλης αυτής της ε, κατάρτισης. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει ε, το πρόγραμμα κατάρτισης, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο μεγάλου εύρους ε, πρόγραμμα κατάρτισης, ίσως να υπάρχει μια δυνατότητα και σε εθνικό επίπεδο να γίνει κάτι. Υπάρχει ανταλλαγή σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή οι δικαστικοί, οι εισαγγελείς, οι νομικοί μπορούν να συμμετάσχουν διασυνοριακά σε προγράμματα σχετικά, ας πούμε και τους υπαλλήλους των δικαστηρίων θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσε ας πούμε ένας Λετωνός υπαλληλός με έναν Ιταλό, με έναν Μαλτέζο, με έναν Γερμανό να μπορούν να ε, συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις. Υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα, έχουν ε, σωματωθεί σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην ε, Λετωνία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτά. Ίσως να σας θέσω και κάποιο άλλο ερώτημα αργότερα. Ευχαριστώ. Thank you for the questions. Um, Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Καταρχάς για τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όπως ξέρετε, έχω πρόσφατα μόνο αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Μπορώ όμως να αντλήσω από την εμπειρία μου για να δώσω κάποιες απαντήσεις. Η δικαστική εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι οργανωμένη με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε αριθμό, γιατί η δομή του όλου συστήματος είναι πιο κεντρική, όμως για παράδειγμα στη δική μου χώρα, τη Φιλανδία, η κατάρτιση είναι κατακαιρματισμένη, είναι διάχυτη αν θέλετε και έτσι δεν βρίσκονται στην στην έκδοση όλα ε, τα δεδομένα. Δεν βρίσκονται στην έκθεση. Επομένως, εν μέρη είναι θέμα δεδομένων. Και εν μέρη ε, δεν έχει ε, αποτυπωθεί σε όλες τις χώρες η ιδέα ότι πρέπει κανείς να το πάρει όλο αυτό το πράγμα από την αρχή και να ξεκινήσει από την αρχή. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά μόνο στη διασυνοριακή ε, κατάρτιση ή εκπαίδευση. Επομένως υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Το να αναμειγνύονται οι άνθρωποι και να έρχονται ε, ε, να, παρακολουθούν κατάρτιση μαζί είναι και ο καλύτερος τρόπος. Αλλά βεβαίως χρειάζονται περισσότερα δεδομένα. Ο Συμπρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Κινίτση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Γιούρη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Λίβε που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και για την παρουσίασή σας. Μας ενημερώσατε για όλο αυτό το έργο που έχει υλοποιηθεί σήμερα στον ε, δικαστικό τομέα και πράγματι είναι αυτό εντυπωσιακό χρειάζεται να μοιραζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ένα πραγματικό χώρο, ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη. Μόλις αναφερθήκατε στις ε, τρομοκρατικές ε, επιθέσεις, στα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν. Υπάρχει ε, η διακίνηση ανθρωπίνων όντων. Υπάρχουν φρικτά φαινόμενα σήμερα και γι' αυτό είναι απαραίτητο οι νομικοί, οι όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου στα κράτη-μέλη, να έχουν κοινή εκπαίδευση. Αυτό είναι εχέγγυο αποτελεσματικότητάς τους. Μετά από τις ερωτήσεις της συναδέλφου, θα ήθελα και εγώ να ξέρω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη. Στη χώρα μου, στην Ιταλία, υπάρχει σχολή δικαστών, βεβαίως, η οποία είναι πολύ σημαντική και χέρι μεγάλου κύρους. Σας ερωτώ όμως, μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και των εθνικών σχολών. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να υπάρχει εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να ασχοληθούν και να αναλάβουν το καθήκον της εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη. Και ε, στη συνέχεια δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις εξελίξεις, να δράσουμε δηλαδή εκ των προτέρων, κυρίως ε, σε επίπεδο νεολαίας, έχοντας άμεση συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με τις ε, νομικές σχολές των χωρών διότι οι νέοι φοιτητέ είναι αυτοί οι οποίοι θα στελεχώσουν τον κλάδο της δικαιοσύνης και έτσι θα μπορέσουν να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Εκ των προτέρων, ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς για τη σωστή και αποτελεσματική εκπαίδευση και τη σύνδεση μεταξύ εθνικών σχολών δικαστών το δίκτυο περί αυτού πρόκειται. Το EGTN ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήδη συνεργάζονται. Επομένως, το σημαντικό είναι οι αρχές που στελεχώνουν τις σχολές δικαστών στα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό να μπορούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για την εκπαίδευση, τη δικαστική. Και άλλωστε και τα πανεπιστήμια υποβάλλουν προτάσεις. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται διασυνοριακά. Ε, από την πείρα μου έχω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου τα πανεπιστήμια, οι νομικές σχολές, να περιλάβουν μαθήματα διδασκαλίας ενωσιακού δικαίου, όχι όμως ως ε, ξεχωριστό δίκαιο, αλλά ως μέρος της ισχύουσας εθνικής ένομης τάξης. Διότι το βασικό είναι να κατανοεί κανείς τις δομές των διαφορετικών αυτών στρωμάτων δικαίου. Ευχαριστώ κύριος Πούντα. Mulțumesc foarte mult, pentru această audiență. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ήθελα να συγχαρώ τη Γενική Διευθύντρια για την ενημέρωση και να της ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Η διαβίου κατάρτιση, η συνεχής κατάρτιση είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερος ε, ε, στο κόσμο της δικαιοσύνης, γιατί λένε ότι αν βρεθούν δύο νομικοί θα δώσουν τρεις διαφορετικές γνώμες. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε κάποια κοινή κατάρτιση. Έχετε κάνει μια αξιολόγηση των δυσκολιών που υπάρχουν σε θέματα εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Συγγνώμη, αλλά μου διέφυγε να τμήμα τη ερώτηση. Είχατε την καλοσύνη να επαναλάβετε. Βεβαίω. Ερωτώ λοιπόν, έγινε μια αξιολόγηση ή λαμβάνεται υπόψη την αξιολόγηση της εφιστάμενης νομοθεσίας που ίσως δημιουργήσει κάποια ε, ε, σύγκρουση συμφερόντων που οδηγεί σε αντιφατικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον γεωργικό προπολογισμό και την πρόσβαση στα γεωργικά κονδύλια. Δεν υπάρχουν μερικές φορές σαφείς ορισμοί για την πρόσβαση αυτή και πολλές φορές ε, είναι δύσκολη η ερμηνεία της ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας γιατί μερικές φορές βρίσκεται στην πηγή των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη εξαιτίας της δυσκολίας ερμηνείας που υπάρχει του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το ερώτημά σας αφορά την βελτίωση της νομοθεσίας. Και στην πατρίδα μου και γενικώ είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη προετοιμασία της κοινοτικής νομοθεσίας, καλύτερη μελέτη επιπτώσεων νομικών κάποιου νομοθετήματος, ώστε να αποφευθούν τέτοιες ε, συγκρούσεις ή τέτοιες δυσκολίες. Αυτό θα πρέπει να το δούμε από την αρχή. Βέβαια τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν πολλές φορές τις ε, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νομικών ή των δικαιικών συστημάτων και οι δικαστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται ε, στο να βρίσκουν την ισορροπία όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Αποτελεί δηλαδή και αυτό το θέμα ένα τμήμα της δικαστικής κατάρτισης. Ευχαριστώ κυρία Κουντρίτσκα. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την ε, Γενική Διευθύντρια για την ενημέρωση που μας έκανε και να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Είπατε ότι καλό θα ήταν και στα πανεπιστήμια, στις νομικές σχολές, ε, ε, να διδάσκεται το ενωσιακό δίκαιο ως συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών, όχι μόνο ως μεμονωμένο μάθημα σε πολλές χώρες ε, και κυρίως στις νέες ε, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ε, για τέτοιες σπουδέ. Αλλά δεν είναι μεγάλος αριθμός των φοιτητών που ενδιαφέρεται. Γιατί ε, το θέμα είναι ότι τέτοιε σπουδέ, τέτοιε κατευθύνσεις δεν επικεντρώνονται μόνο στην ιεράρχηση του, ε, του κοινοτικού δικαίου, συνθήκες πρωτογενές παράγω και ούτε καθεξής. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον ε, όλοι οι επαγγελματίες στον τομέα της ε, δικαιοσύνης ε, αλλά και οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα και την ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μόνο τον τρόπο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Γιατί αν ο κόσμος, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταλαβαίνουν την γεωργική νομοθεσία, την νομοθεσία για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία του καταναλωτή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις πολιτικές, ε, η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στις πολιτικές αυτές θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Γιατί θα επαφίεται περισσότερο στην ερμηνεία τους και άρα θα είναι διαφοροποιημένη. Οπότε θα πρότεινα να αξιοποιήσουμε τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα που έχουν και πανεπιστημιακό και διδακτικό έργο και επικεντρώνονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημόσιας Διοίκησης που εδρεύει στην Ευρω... στις Βρυξέλλες ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Δι... Επιστήμης. Να αξιοποιήσουμε και αυτά τα Ινστιτούτα και αυτούς τους θεσμούς γιατί είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι μόνο το ενωσιακό δίκτυο, δίκαιο. Τότε μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι οι ασκόντες νομικά επαγγέλματα καταλαβαίνουν πλήρως το ενωσιακό δίκαιο που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν, έχοντας καλύτερη γνώση και των ευρωπαϊκών πολιτικών σε προγενέστερο επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο σχόλια. Καταρχήν, η νομική κατάρτιση σε επίπεδο νομικών σχολών, πανεπιστημίων ε, θα αφορά μαθήματα που δίνουν μια γενική εικόνα της νομοθεσίας. Και μετά έχουμε τη ένομη τάξη κάθε χώρας ε, μέλους. Αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να διδάσκεται στους επιμέρους τομείς, ώστε να γίνεται αντιληπτό ε, και το θέμα της πολιτικής και το θέμα της νομοθεσίας. Αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει οι δικηγόροι να γνωρίζουν περισσότερο για την πολιτική, ε, τις πολιτικές ε, και την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, γιατί οι δικηγόροι δεν θα πρέπει να είναι απλοί τεχνοκράτες που θα εφαρμόζουν ή θα ερμηνεύουν συσταλτικά ε, συγκεκριμένες ε, νομοθετικές ρήτρε ή συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Θα πρέπει να έχουν μια ευρύτερη αντίληψη και κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σκέλος και τμήμα όλων των νομικών καταρτήσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Διευθυντρία για την επιτυχία που είχαμε σε θέματα κατάρτισης δικαστικών και να τονίσω την ερώτηση της κυρίας Τσινίτση για το ρόλο των πανεπιστημίων και των νομικών σχολών. Έχω μία ερώτηση. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για χρηματοδότηση της ε, συνεργασίας των ε, καθηγητών ε, των νομικών σχολών, για παράδειγμα. Ή υπάρχουν κοινά προγράμματα σπουδών σε κάποια πανεπιστήμια χωρών μελών. Thank you very much for the question. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Αυτά τα κονδύλια δεν μπορούν να δοθούν για τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο, αλλά το πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει τμήμα μιας ομάδας, ας πούμε, που ζητά κονδύλια για τους καθηγητές νομικής. Δεν μπορούν να ζητήσουν όμως ε, ε, κονδύλια για τη διδασκαλία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Κιώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός και βεβαίως πρέπει να τον ενισχύσουμε, την κατάρτιση και την περαιτέρω κατάρτιση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα θέματα της περαιτέρω κατάρτισης που σας απασχολούν για τον τομέα αυτό. Και επίσης υπάρχει κάποιο είδους αξιολόγηση αυτών των συνολικών προγραμμάτων κατάρτισης και υπάρχει ίσως και μια εσωτερική ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών από την οποία θα μπορούσαμε ίσως να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα. Αν δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνουμε έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, έχουν τα αποτελέσματα που τελικά περιμέναμε. Καταρχάς, να πω ότι ο μηχανισμός που υπάρχει, υπάρχει για να βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Στην παρούσα φάση επικεντρωνόμαστε κυρίως στο ποσοτικό, στην ποσοτική πτυχή. Βεβαίως η ποιοτική πτυχή είναι πάντα δύσκολο να μετρηθεί, αλλά όταν αξιολογούνται τα αποτελέσματα για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης, εκεί τότε ναι γίνονται και γίνεται αξιολόγηση και κάποιων ε, ποιοτικών δικτών. Όπως είπα, στην πρώτη γραμμή της κατάρτισης έχουν μπει οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Ε, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε και με τους ε, δικαστικούς κλητήρες και με τους υπαλλήλους των δικαστηρίων. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάρτιση των νέων δικηγόρων, γιατί είναι σημαντικό από την αρχή, όχι μόνο των δικηγόρων, αλλά και των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, από την αρχή της εξάσκησης του επαγγελματό τους να μπορούν να κατανοήσουν όλη τη δομή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την νομική κουλτούρα. Τώρα, σε αφορά τα θέματα είναι αρκετά ευρύ το φάσμα αυτό. Όπως είπα υπάρχουν θέματα αστικού δικαίου, υπάρχουν θέματα ποινικού δικαίου, εμπορικό δίκαιο, ε, ουσιαστικό ποινικό, θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα διδασκαλίας αυτό γιατί σχετίζεται άμεσα ουσιαστικά με κάθε θέμα, με κάθε ε, πρόβλημα που μπορεί να προκύψει και μετά οι νέε τάσεις επίση που υπάρχουν ε, και που προκύπτουν ε, μετά από τα τραγικά συμβάντα στην Ευρώπη. Ε, αντιμετώπιση του, της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους για να αναγνωρίζουν τι συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο διαχειρίζονται, έτσι ώστε να κατανοούν ας πούμε, οι δικαστές τι είδους υπόθεση είναι αυτή η υπόθεση που πρέπει να δικάσουν. Ας πούμε, για τους δικαστικούς είναι καλό να γνωρίζουν τι είδους ποινή θα ήταν καλό να επιβληθεί. Είναι σωστό να στείλουμε κάποιον στη φυλακή που μπορεί να παστικοποιηθεί ακόμη περισσότερο ή είναι καλύτερο να του αποδώσουμε μια διαφορετική ποινή ώστε να μπορέσουμε να τον ενσωματώσουμε και πάλι. Οπότε ως προς αυτό υπάρχει ένας νέος ε, ανεξερεύνητος τομέας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Σα άκουσα κυρία μου με μεγάλη προσοχή και εκτίμησα ιδιαίτερω την πρόταση που εκφέρατε. Οι νομικοί δεν είναι τεχνοκράτες και πρέπει να το υπενθυμίσουμε πράγματι. Γιατί οι νομικά επαγγέλματα δεν βρίσκονται εδώ για να εφαρμόσουν τεχνικούς κανόνες αλλά και να εκτιμήσουν το διακύβευμα στην κοινωνία. Και κάθε φορά που γίνεται αναφορά στο ρόλο των πανεπιστημίων θα πρέπει να τονίσουμε το ισχυρό του σημείο ότι δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν περιορίζονται στην τεχνική διδασκαλία στη Γαλλία. Ο καθηγητής Μισελ Κλαπιέ έχει δημοσιεύσει ένα φανταστικό έργο με τίτλο το ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα και η ανάλυση του δεν περιορίζεται στην περιγραφή των θεσμικών οργάνων. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι μιλούμε σήμερα για εκπαίδευση δικαστική και πολύ φοβούμαι ότι θα την περιορίσουμε μόνο στην κατάρτιση, δηλαδή στην τεχνική εκπαίδευση μόνο. Ε, σαφέστατα πρέπει κανείς να γνωρίζει το ενωσιακό δίκαιο και πρέπει να γνωρίζουν και το δίκαιο των βασικών χωρών. Όμως, όταν μιλούμε για μια κουλτούρα ενωσιακού δικαίου, αυτό με ανησυχεί κάπως και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Εγώ είμαι Γάλλος και θεωρώ ότι ε, είναι μια έννοια γερμανικής προέλευσης η οποία δεν έχει ε, αποκτήσει πραγματικές ρίζες στη Γαλλία ε, και είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους φοιτητές μας, γιατί εμείς μιλούμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη ε, είναι μια έννοια γαλλική από το 1789 και δεν ταυτίζονται με τον όρο θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι λεκτική διαφορά μόνο. Ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου βασίζονται τη συμφιλίωση μεταξύ της ατομικής θεωρίας και της συνολικής και ολιστικής προσέγγισης. Όλα αυτά τα έχει αναλύσει πολύ επιτυχημένα ο Λουκ Φερή. Επομένως, ε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο καθένας έχει τη δική του νομική παράδοση και θα πρέπει το άνοιγμα προς τους άλλους να γίνεται και να συμφιλιώνονται με την ε, διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής παράδοσης στην ένωμη τάξη. Αυτή είναι η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι εδώ ακριβώς συζητούμε για το ότι μοιραζόμαστε εμπειρίες. Πράγματι, η εκπαίδευση που δίδεται στους ασκόντες νομικά επαγγέλματα ε, δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως, έχει να κάνει και με δικαστικά ζητήματα σε ευρύτερο πεδίο και με ευρύτερες δεξιότητες. Το να μοιραζόμαστε εμπειρίες, βιώματα, είναι το διασυνοριακό στοιχείο της εκπαίδευσης αυτής με σκοπό ακριβώς να λύσουμε αυτά που αναφέρατε. Ξέρετε, στη νομική γλώσσα χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις για διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές λέξεις μερικές φορές για το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό οι δικηγόροι να το κατανοούν αυτό για να μην τις χρησιμοποιούν μηχανικά, αλλά για να ξέρουν τι κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Ελπίζω επομένως ότι με τη διασυνοριακή εκπαίδευση θα μπορέσουμε να λύσουμε και να δουλέψουμε πάνω στα ζητήματα που υπάρχουν και που αναφέρατε πράγματι. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν θέλει κάποιος άλλος να θέσει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά, ε, κυρία Άστολα, για το ότι ήρθατε σήμερα μαζί μας εδώ ε, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο συμπρόεδρος κύριος Μωράης έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ε, να σας εκφράσω τις ευχαριστίες ε, τις δικές μου προσωπικά αλλά και των λοιπόν συναδέλφων από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών απαντήσατε σε ερώτηση για ποινικού δικαίου και να σας πω ότι πολλά μέλη της Επιτροπής μας ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και ε, ας νομοθετούν ε, πάνω σε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης των δικαστών στα ποινικά δικαστήρια είναι ένα ζήτημα πρακτικό που μας απασχολεί καθημερινά. Μας διαφωτίσατε και χρειαζόμαστε τη συνεργασία με εσάς και με την Επιτροπή Γιούρη για τα θέματα αυτά. Καλή επιτυχία στο έργο σας και ευχαριστώ και, στα, και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που ήρθαν σήμερα σε αυτή τη κοινή συνεδρίαση.